Colleghi, riprendiamo la seduta. Αρχίζει η συνεδρίασή μας. Ο κύριος Γιακολίνο θα μας μιλήσει για την τελική του έκθεση. Έχει 20 λεπτά για να μας επεξηγήσει την τελική έκθεση και μετά θα λάβουν το λόγο οι εισηγητές οι συντονιστές με συγχωρείτε. Κύριε Γιακολίνο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Όπως ξέρετε την προηγούμενη εβδομάδα ενεκρίθη η ενδιάμεση, ενδιάμεση έκθεση, κάτι το οποίο κατοχύρωσε τις καλές προθέσεις όλων που αποτελεί σημείο εκκίνησης. Συζητήθηκε το θέμα την Τρίτη στο Στρασβούργο, ενεκρίθη λοιπόν η ενδιάμεση έκθεση. Στις 30 Μαΐου υπέβαλα το τελικό κείμενο. Προσπάθησα να μειώσω τον όγκο αποσύροντας ε, επικαλύψεις, θεωρώντας ότι το τελικό προϊόν θα πρέπει να είναι ευέλικτο και καθόλου ογκώδες για να είναι ευανάγνωστο. Υπενθυμίζω τις 744 τροπολογίες που είχαμε αρχικά στην ε, ενδιάμεση έκθεση Είχαμε πολυάριθμες τροπολογίες και στο, κατά τη συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα, την Τρίτη, στην Ολομέλεια. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε το καλύτερο δυνατό κείμενο μέσα στα πλαίσια της ενδιάμεσης έκθεσης και επί της ουσίας ότι απετέλεσε αντικείμενο έγκρισης της ενδιάμεσης έκθεσης, αν και δεν συμπεριληφθεί στην τελική έκθεση, είναι αναπόσπαστα, αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής έκθεσης, όπως θα διαμορφωθεί. Προσπαθήσαμε να προσθέσουμε ορισμένα καινοτόμα στοιχεία είχαμε να κάνουμε με έναν μεγάλο όγκο εργασίας μέσα στα πλαίσια των, και των ακροάσεων και στόχος της έκθεσης είναι να ορίσουμε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και του ξεπλήματος του βρώμικου χρήματος μέσα στα πλαίσια μιας ενιαίας νομικής ε, βάσης στα κρατη με αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων. Αυτό αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ε, δικαστικής συνεργασίας. Επίσης, να δούμε ποιες επιχειρήσεις έχουν καταδικαστεί για να υπάρχει αποκλισμός τους από τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαγωνισμό. Πρόκειται για τις επιχειρήσεις που έχουν σπηλωθεί γιατί πρόθεσαν παράνομες δραστηριότητες σε συνεργασία με το δημόσιο τομέα. Έχουμε και τις μαύρες λίστες των επιχειρήσεων αυτών που δεν θα πρέπει να έχουν καμία σχέση με, τις δημόσιες, με το δημόσιο των κρατών μελών, με το δημόσιο τομέα. Επίσης μας ενδιαφέρει η αντιμετώπιση των εγκλημάτων, του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο με βάση τα πρόσφατα επεισόδια που γνωρίσαμε κάτι το οποίο έχω αναφέρει μέσα στα πλαίσια της διερεύνησης της όλης διαδικασίας. Επίσης, μας απασχόλησε η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, αλλά και με τρίτες χώρες μας απασχόλησαν θέματα κατασχέσεων και δημεύσεων και βρισκόμαστε σε μια φάση διαπραγμάτευσης μεταξύ θεσμικών οργάνων. Το φάκελο για τις ε, κατασχέσεις τον είδαμε ήδη μέσα στα πλαίσια του αστικού και του ποινικού δικαίου. Τώρα μας ενδιαφέρει και η ανιχνευσιμότητα των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, συνεργασία με εμπορικά επιμελητήρια και συμβολεογράφους, θέματα που σχετίζονται με τους φορολογικούς παραδείσους. Έγινε λόγος στην Ιλλανδία για τις προαπαιτήσεις που χρειάζονται για την άρση του τραπεζικού απορρίτου μέσα στα πλαίσια και των φορολογικών παραδείσων. Αυτό εμείς το εγκρίναμε και στην τελική έκθεση. Πιστεύουμε ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι πιο σωστή, πιο δίκαιη και να δρά άμεσα. Θεωρήσαμε ότι ως προς το ξέπλυμα θα πρέπει να έχουμε σαφείς ενδείξεις για την ανείχνευση του πραγματικού δικαιούχου της συναλλαγής. Και επίσης θεωρήσαμε ότι σε αυτή τη φάση θα πρέπει να επισύρουμε την προσοχή στα παράνομα στοιχήματα, στους παραδείσους αυτούς, ιδιαίτερα στην Ασία. Διότι επηρεάζουν την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο. Το οργανωμένο έγκλημα έχει παγκόσμια διάσταση και γι' αυτό χρειάζεται και μία πραγματική ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να δρουν ισότιμα στα κράτη-μέλη και να μην υπάρχει ούτε φοροδιαφυγή ούτε φοροαποφυγή. Τις τελευταίες μέρες λάβαμε ανησυχητικά στοιχεία για το κόστος της φοροδιαφύγης στην Ευρώπη. Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, ε, Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ σας αναφέρομαι στις ε, σημαντικότερες χώρες που πλήττονται γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η φοροαποφυγή σημαίνει απώλεια χρημάτων από το δημόσιο κορβανά. Γι' αυτό θα πρέπει τα κράτη να μπορούν να παρέμβουν αμεσότερα στον τομέα της, να μπορούν να παρέμβουν στον τομέα της πρόνοιας, της υγείας και της ε, υπεράσπισης των πλέον ευάλωτων κατηγοριών με βάση την καλπάζουσα φτώχεια που διακρίνει την ιστορική αυτή στιγμή της ευρωπαϊκές χώρες. Θέλουμε να ορίσουμε το οργανωμένο έγκλημα, να υπάρχει μία σωστή οριοθέτηση, όπως επιθυμούν και οι πολιτικές ομάδες. Συνεργαστήκαμε με τους σκιώδεις και με τους συντονιστές για να ορίσουμε ένα κείμενο το οποίο να είναι κατανοητό. Προσπαθήσαμε να οριοθετήσουμε καλύτερα αυτή την εργασία, μειώνοντας τον όγκο του κειμένου, χωρίς να πλήξουμε το περιεχόμενο μέσα στα πλαίσια αυτής της ε, γενικής ε, πρόβλεψης, διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το τελικό κείμενο, το οποίο να περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα της ενδιάμεσης έκθεσης. Σε αυτή τη φάση λοιπόν συγκεφαλαίωσης θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφής ε, ως προς τις οικονομικές δραστηριότητες. Μας ενδιαφέρει και ο ρόλος του Ευρωπαίου εισαγγελέα για να είναι ουσιώδης οι έρευνες. Μιλάμε λοιπόν για συγκεκριμένα και αποτελεσματικά κείμενα για τους συνεργάτες ε, στη δικαιοσύνη και τους μάρτυρες καταβάλαμε κάθε προσπάθεια γιατί το κείμενο αφορά το οργανωμένο έγκλημα και την δουλεμπορία. Προσπαθήσαμε να συγκεφαλαιώσουμε τα δεδομένα, τα στοιχεία που μας έδωσαν οι πολιτικές ομάδες. Ορίσαμε ένα σύστημα το οποίο ε, μιλά για τις συγκληματικές οργανώσεις και τη δραστηριότητά τους στην πραγματική οικονομία. Μιλήσαμε για την επαναχρησιμοποίηση των ε, κατασχεθέντων και αντιμετώπιση των ε, καταδικασθέντων σε, για αδικήματα που δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Θεωρούμε λοιπόν ότι χρειάζεται μία νέα διάσταση, μία νέα προσέγγιση και θεωρώ ότι η εργασία αυτή ολοκληρώθηκε με μία ας πούμε ενωσιακή προσέγγιση και χωρίς διαφορές. Θεωρώ, Πρόεδρε, ότι εδώ θα πρέπει να σταματήσω δεν χρησιμοποίησα το χρόνο που μου διαθέσατε, διότι τα θέματα αυτά έχουν πολύ καλυφθεί από την ενδιάμεση έκθεση, η οποία εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ε, είτε υποδείξεις υπενθυμίζοντας ότι αυτό που μετράει είναι η καλή εργασία αυτής της Επιτροπής που εξαρτάται από τον αριθμό των συναδέλφων που συνεισφέρουν. Κατά την ε, κατάρτιση των, κατάρτιση ε, των τροπολογιών Είδαμε ότι ήταν ε, πάρα πολλές και από πολλούς. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία είναι να υποβάλλονται και από συναδέλφους ε, οι οποίοι παρευρίσκονται συχνά στις εργασίες μας. Από την ε, καρποφόρα αυτή η συνεργασία πιστεύω ότι ότι θα υπάρξουν και βελτιώσεις. Φτάσαμε σε 77 τροπολογίες συμβιβασμού, οι οποίες ε, καταρτίστηκαν και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή, μειώνοντας τον αρχικό αριθμό. Μιλάμε για τις τροπολογίες, οι οποίες ήταν απολύτως αναγκαίες για να βελτιώσουμε το κείμενο το οποίο εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Νοβίτα. Υπάρχουν ορισμένα νέα στοιχεία στην τελική έκθεση, τα οποία σας έθεσα υπόψη. Ευχαριστούμε πολύ. Αρχίζει η συζήτηση. Το λόγο έχει ο κύριος Κίρκοπ. Thank you Ευχαριστώ και με συγχωρείτε που άργησα για την παρουσίαση του κυρίου Γιακολίνο. Θα ήθελα και πάλι να τον συγχαρώ για τα όσα έκανε, για τον τρόπο με τον οποίο τα έκανε. Η ομάδα μου δεν μπορεί να συμφωνήσει με τα πάντα, το γνωρίζει είχαμε στην ενδιάμεση έκθεση και τα συμπεράσματα τα οποία επέστηραν την προσοχή μας πάνω σε ορισμένα πράγματα τα οποία είναι απολύτως σωστά και χαίρομαι γι' αυτό. Θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια πάρα πολύ σύντομα σχετικά με τα θέματα που παρουσίασε πριν από λίγα λεπτά σε σχέση με το θέμα των φόρων, της φοροδιαφυγής. Είναι ένα θέμα που όπως γνωρίζει συζητείται έως είναι στο G8 στη Σύνοδο Κορυφής η οποία συνεδριάζει τις τελευταίες μέρες στην Βόρεια Ιρλανδία υπό την Προεδρία του Ηνωμένου Βασιλείου. Το θέμα αυτό συζητείται. Εγώ μιλώντας ως επαγγελματίας, διότι είμαι δικηγόρος, είχα πάντοτε ε, μια άποψη για τους φόρους ε, υπήρχε πάντοτε μια διαφορά ανάμεσα στα άτομα τα οποία αποφεύγουν την πληρωμή που είναι υποχρέωση νομική και αυτή που αποφεύγουν την φορολόγηση ή τακτοποιούν τα πράγματα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειάζεται να πληρώσουν ε, περισσότερους φόρους από ό,τι θα ήσαν υποχρεωμένοι με τα περιουσιακά του στοιχεία. Όλο όσο περνάει ο χρόνος βρίσκουμε ότι οι πολιτικοί ηγέτες στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο συμπεραίνουν ότι ακόμη και τα άτομα που αποφεύγουν να ε, πληρώσουν ε, τους φόρους σε σχέση με τους παράνομους πρέπει να ελέγχονται, να τους υπενθυμίζει κανείς τις ευθύνες τους, τις ηθικές και άλλες. Υπάρχει τώρα μεγάλη συνεργασία σε ολόκληρο τον κόσμο ε, που τους προτείνει να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις τους αυτοί προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν τους φόρους τους. Δεν υπάρχει βεβαίως τίποτα το παράνομο σε αυτό. Θέλουμε ε, να υπάρξει συνεργασία και να παροτρύνουμε ε, τα άτομα να επενδύουν στις χώρες μας. Αλλά αυτό θα πρέπει ε, να το ξεδιαλύνουμε, να το διευκρινίσουμε. Αυτό ε, το κάνετε στην έκθεσή σας κύριε Γιακολίνα, υπενθυμίζετε στα άτομα ότι εκτός από αυτό το θέμα της φόρα αποφυγής και τους νόμους που ισχύουν στις διάφορες χώρες υπάρχει επίσης ε, μεγάλη εγκληματικότητα η οποία συνεχίζεται σε σχέση με τα θέματα αυτά. Η αποφυγή βεβαίως είναι μια οικειοθελής πράξη, αλλά η εγκληματικότητα που συνδέεται με αυτήν είναι ουσιαστική, όχι μόνο προς το ύψος των ποσών που εμπλέκονται, που είναι δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, αλλά επίσης και ε, σχετίζεται με άλλα πράγματα που συνδέονται με τα χρήματα αυτά ή με το γεγονός ότι το φορολογικό σύστημα δεν λαμβάνει υπόψη τα ποσά αυτά. Υπάρχουν και άλλα εγκλήματα και αδικήματα ε, στην Ευρώπη. Καμιά φορά η χρηματοδότηση βιαίων εγκλημάτων, καμιά φορά τα χρήματα αυτά πηγαίνουν στα χέρια αυτών που οργανώνουν και εκτελούν τρομοκρατικές πράξεις κατά των πολιτών μας. Το θέμα είναι βεβαίως ότι οι άνθρωποι πρέπει να πληρώνουν περισσότερους φόρους ή να πληρώνουν τους φόρους που οφείλουν να πληρώνουν αυτό το, το ποσό, το επίπεδο ε, ε, χρημάτων είναι τόσο μεγάλο, τόσο υψηλό, ώστε αν θέλετε παροτρύνει την εγκληματικότητα και ασχολούμεθα εδώ με σοβαρά δικήματα, με τρομοκρατία, την χρηματοδότηση που υπάρχει, τη χρηματοδότηση αυτών των εγκληματικών πράξεων, πώς τα χρήματα διοχετεύονται, το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, όλα αυτά τα πράγματα τελικά τα θέματα τα οποία αναφέρατε κύριε Γιακολίνο στην έκθεση αυτή και στον τομέα αυτό είναι τόσο σημαντικά για όλους μας ώστε χρειάζεται ε, να εμβαθύνουμε περισσότερο στα θέματα αυτά, ίσως να το κάνουμε στην τελική έκθεση ή ε, ως μια άλλη, έναν άλλο υποκλάδο, υποτομέα της εργασίας μας, διότι χωρίς τα χρήματα, χωρίς τους πόρους, αυτούς το έγκλημα θα είναι πολύ πιο περιορισμένο και θα περιοριστούν οι δυνατότητες της αποτελεσματικής τρομοκρατίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κύρκοπ. Η κυρία Φεγιόμ. Ναι. ναι. Θα ήθελα επίσης πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Σαλβατόρε για την προσπάθεια που κατέβαλε για να εκπονήσει αυτήν την έκθεση. Νομίζω ότι το τελευταίο έτος της εντολής μας, της θητείας μας μετά από πολλές ακροάσεις, αφού συνομιλήσαμε με εμπειρογνώμανες, κάναμε πολλά και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχανε σε αυτήν την προσπάθεια συνεργασίας. Στο παρελθόν χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε επίσης κάποια προβλήματα οι συναδελφοί μας δεν ήταν ε, πάντοτε ε, στις ακροάσεις ε, και αυτό αναφέρθηκε στις τροπολογίες της ενδιάμεσης έκθεσης. Πολλά από αυτά που συμφωνήσαμε έχουν περιληφθεί τώρα στην έκθεση και πρόκειται για τροπολογίες τόσο από τη δική μου πλευρά όσο και από άλλες ομάδες. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω όλους. Εδώ σε αυτή την εποχή όπου υπάρχει όλο και λιγότερη εμπιστοσύνη στην πολιτική, στους θεσμούς, νομίζω ότι είναι ζωτική σημασία να συζητούμε για να δούμε πώς τα χρήματα, τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δαπανώνται από τα κράτη-μέλη και από άτομα. Είναι ζωτική σημασίας να κάνουμε συστάσεις για όλους που ασχολήθηκαν με την διαφθορά στα δικαστήρια θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, να καθαρίσουμε ε, το δικό μας ε, σπίτι προτού αποκτήσουμε την εμπιστοσύνη των ε, πολιτών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αρχίσει διαδικασίες εργασίες ε, σχετικά με το γραφείο του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα, διότι αυτό θα είναι ένα βήμα θετικό επίσης ε, και τα, για τα ε, εθνικά γραφεία εισαγγελέων. Αυτά είναι συγκεκριμένα μέτρα που μπορούμε να συστήσουμε. Επίσης ανησυχώ διότι δεν ξέρω αν τα κράτη-μέλη θα ακολουθήσουν τις συστάσεις. Αν εξετάσουμε ε, την έκθεση για την φορολογική ε, φοροδιαφυγή που υιοθετήθηκε στην Ολομέλεια, μόνο ε, μερικές από τις συστάσεις μας, ένα μικρό ποσοστό συστάσεων έγινε δεκτό από το Συμβούλιο. Ελπίζω στο τέλος της θητείας μας ότι θα έχουμε ένα σαφές μήνυμα του ποιες είναι οι συστάσεις μας, το πώς μπορεί να βελτιώσουν την κατάσταση ε, τα κράτη-μέλη, ε, δαμάζοντας ε, την, την φοροδιαφυγή, την διαφθορά. Ε, δεν πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο, αλλά παγκόσμιο φαινόμενο και σε εποχή οικονομικής κρίσης πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε μερικά από τα στοιχεία της έκθεσης. Η έκθεση αυτή δεν είναι και τόσο διαφορετική από την ενδιάμεση ε, έκθεση. Σε μερικά σημεία είναι ε, και συντομότερη. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση. Παρέντος χάρη το τμήμα που αναφέρεται στη μάφια. Δεν υπάρχει εκεί πάρα πολύ περιεχόμενο. Γιατί, γιατί μικρίναμε αυτήν, αυτήν, αυτό το τμήμα σε σχέση με την ενδιάμεση έκθεση. Άλλα δύο στοιχεία για τα οποία θα ήθελα να εκφράσω σχόλια. Πρώτον, το 18, το σημείο 18 στην σελίδα 17, ε, στην δική μου γλωσσική εκδοχή όταν μιλάτε για την Eurojust και την Europol, λέτε ότι θα ήταν καλό να χρησιμοποιούμε διαδικτυακές πληροφορίες. Οι Ευρωπαίοι είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι όσον αφορά στα στοιχεία αυτά και στα δεδομένα αυτό. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις σας όταν ε, μιλάτε ε, για τους οργανισμούς ε, του διαδικτύου. Δηλαδή να δίνονται πληροφορίες όταν πρόκειται για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς, του ξεπλήματος μαύρου χρήματος ή θα έπρεπε ίσως να βελτιώσουμε κάπως τη διατύπωση. Και μετά το σημείο Y, το οποίο σχετίζεται ε, με την, ε, τα νόμιμα παιχνίδια, νόμιμα παιχνίδια, όχι παράνομα, τα οποία λέτε ότι πρέπει να υποστηριχθούν, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν είναι αυτή η καλύτερη ιδέα, διότι τα παιχνίδια δεν είναι πάντοτε νόμιμα σε όλες ε, τις χώρες μέλη. Θα ήθελα ακόμη ε, μερικές ε, λεπτομέρειες, μερικές διευκρινήσεις ε, για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν μερικά νέα στοιχεία, αλλά νομίζω ότι σε αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα θα μπορέσετε να βελτιώσετε την έκθεση και ελπίζω ότι θα μπορούμε να μεταδώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα στους πολίτες μας. Ο κύριος Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερο και τον εισηγητή για την πολύ και δύσκολη δουλειά που έκανε καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλει. Ωστόσο, έχω να επισημάνω μια διαδικασία, μάλλον μια λεπτομέρεια διαδικαστική. Είπε κάτι και ο συγγετής, και αυτός να το πρόσεξε. Από τη δική μας πολιτική ομάδα εμείς δεν καταθέσαμε τροπολογίες ούτε άλλωστε για την Ολομέλεια, για την ε, Σύνοδο του Στρασβούργου. Γιατί εμείς απέσχομεν στην τελική ψηφοφορία. Γιατί θεωρήσαμε ότι ήταν πολύ περιορισμένος ο χρόνος της συζητήσεως και θεωρήσαμε ότι δεν ήταν ενδεδειγμένο να καταθέσουμε έναν μεγάλο αριθμό τροπολογιών αλλά θεωρήσαμε επίσης ότι οι τροπολογίες που θα θέλαμε να καταθέσουμε θα έπρεπε να κατατεθούν για την τελική έκθεση. Γι' αυτό τηρήσαμε άλλωστε και τη στάση που εξήγησα στην ε, ψηφοφορία. Χρειαζόμαστε βέβαια χρόνο. Αλλά να δούμε μήπως μπορούμε να ακολουθήσουμε άλλη διαδικασία η πολιτική μας ομάδα βλέπει το πρόβλημα ότι και ίσως να καταθέσουν και άλλες ομάδες πολλές τροπολογίες να εξετάσει το ενδεχόμενο ο εισηγητής μήπως στο τελικό του κείμενο διατυπώσει πιο συγκεκριμένα συμπεράσματα στα οποία να περιλάβει συστάσεις με στόχο να εξασφαλιστεί ότι το όλο θα παραμείνει ορατό και ότι θα αφήσει κάποιο ίχνος. Γιατί πρόκειται για ένα κείμενο, για ένα θέμα το οποίο θα παίξει σημαντικό ρόλο και στον προεκλογικό αγώνα. Λοιπόν αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ίσως αξίζει να σκεφτεί ο συγκητής και ξαναλέω ότι ένας αριθμός τροπολογιών τις οποίες δεν καταθέσαμε για την διάμεση έκθεση θα κατατεθεί τώρα για την τελική. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άλμπρεχτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή για το έργο που επετέλεσε. Εξετάζοντας το σχέδιο της τελικής εκθέσεως, πρώτα πρώτα επισημαίνω ότι είναι πολύ εκτεταμένο το είχα δει αυτό και στο κείμενο της ενδιάμεσης έκθεσης και εν τέλει κάπως είναι ασαφές ποια είναι τα συγκεκριμένα συμπεράσματα τα οποία αντλούμε από τις εργασίες της παρούσας Επιτροπής. Δηλαδή τελικά τι εντολή δίνουμε στον νομοθέτη, άρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στον εαυτό μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ποια είναι η σχέση με τα μέτρα τα οποία συζητούμε. Δηλαδή, εάν ρίξετε μια ματιά στις εργασίες της Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών, όπου εκπονούνται οδηγίες για το πλήσιμο του παράνομου χρήματος, για την καταπολέμηση των απατών, για την καταπολέμηση απατών σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, βεβαίως και με κατασχέσεις, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρα τα όσα έχουν τεθεί τώρα εδώ επιτάπητος ως θέματα. Και ετήθηκε το ερώτημα Πώς θα εξασφαλίσουμε ώστε τα όσα θα περιλάβουμε εδώ στην τελική έκθεση θα υποστηριχτούν και ουσιαστικά από όλους και όλες εδώ στο Κοινοβούλιο και από τις άλλες δηλαδή κοινοβουλευτικές επιτροπές. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι αρκετά συγκεκριμένα. Δηλαδή, αν δεν είναι συγκεκριμένες οι αξιώσεις μας, τότε πιο πολλοί θα θυμηθούν τον τρόπο με τον οποίο συζητούμε εδώ, τις αντιπαραθέσεις, γιατί για μένα δεν είναι σαφές πώς θα προχωρήσει το θέμα αυτό. Θα προχωρήσουμε όπως μέχρι τώρα. Αυτό για μένα μου φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο ενδεδειγμένο. Επαναλαμβάνω ότι δεν είναι αρκετά συγκεκριμένα τα συμπεράσματα. Ίσως πρέπει λοιπόν να περιοριστεί ο εισηγητής σε λίγες παραγράφους χωρίς να επαναλάβει όλο τον αριθμό ενδεχομένων εναλλακτικών επιλογών, δυνατοτήτων κτλ. Είναι σαν ένα μεγάλο μπουκέτο αυτή τη στιγμή αυτό που μας προσφέρει και εμένα με καθιστά κάπως επιφυλακτικό. Και ένα θέμα που απασχολεί εμάς της ομάδας των πράσινων δηλαδή και που θεωρούμε ότι δεν έχει περιληφθεί επαρκώς. Εξακολουθώ να πιστεύω ακράδαντα ότι η εναρμόνιση διαδικαστικών προτύπων, για παράδειγμα για τη συνεργασία αστυνομικών και δικαστικών αρχών, ότι αυτή πρέπει να είναι βασική προϋπόθεση για την βελτίωση της συνεργασίας. Επίσης, η εναρμόνιση βασικών αρχών του ποινικού δικαίου, του συνταγματικού δικαίου, των διαφόρων θεμελιωδών δικαιωμάτων, είναι απόλυτα σημαντικά και επίσης αποτελούν το θεμέλιο της βελτίωσης της συνεργασίας. Αυτά όμως περιλαμβάνονται πολύ περιορισμένα εδώ. Λέμε για παράδειγμα ότι θέλουμε να προωθηθεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την διεξαγωγή ε, των ανακρίσεων. Αυτό χρειάζεται αμοιβή αναγνώριση. Δεν δημιουργεί όμως κοινά πρότυπα. Το μόνο που κάνει ίσως είναι να φτιάχνει μια καταφαντασία εμπιστοσύνη στις ε, οικίες δικονομίες, αλλά δεν δίνει μια συγκεκριμένη βάση για συνεργασία. Επίσης έχουμε πολύ περιορισμένο αριθμό μικτών ομάδων ερευνών ή ανακρίσεων μεταξύ δηλαδή διαφόρων χωρών μελών. Και αυτό δεν γίνεται διότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο ισότιμο των δικαιικών αρχών, των δικαιικών συστημάτων. Αυτά πρέπει να αποκατασταθούν. Δυστυχώς ελείπει εντελώς, σχεδόν εντελώς αυτό το μέρος από την έκθεση. Το τονίσαμε αυτό ως πράσινη και θα επιμείνω και θα επιμείνουμε ότι χρειάζεται εναρμόνιση των διαδικαστικών αρχών, των αρχών δηλαδή των διαδικασιών. Δεν θέλουμε να περιοριστούν προς Θεού οι έρευνες Θέλουμε να υπάρξει ένα κοινό θεμέλιο πάνω στο οποίο να μπορούν να συνεργαστούν οι αρχές, να υπάρξει αμοιβαία εμπιστοσύνη στις διάφορες διαδικασίες και όλες οι άλλες συμπαθητικές αξιώσεις που περιλαμβάνει το κείμενο, αυτά είναι όλα γνωστά λίγο πολύ, τα θέλουμε, αλλά είναι ευχολόγιο. Όλοι τα λένε αυτά. Αλλά ο δρόμος που θα οδηγήσει στην εκπλήρωση αυτή του ευχολογίου δεν είναι, ξεκάθαρος. Γι' αυτό θεωρώ ότι ως και κοινοβούλιο πρέπει να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα, να πούμε ότι θέλουμε την εναρμόνιση ορισμένων προτύπων, για παράδειγμα, για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, όπου θεωρώ ότι η ανάγκη αυτή είναι προφανής. Κοινοί κανόνες είναι το α και το ω. Μόνο τότε, εφόσον υπάρξουν αυτοί δηλαδή, θα βελτιωθεί η συνεργασία. Ευχαριστούμε uh, uh, uh, Ευχαριστώ και ευχαριστώ τον Σαλβατόρε Γιακολίνο. Η θέση του ήταν παράλογη, δηλαδή έπρεπε να υποβάλει την τελική έκθεση πριν ψηφίσουμε την ενδιάμεση. Άρα έπρεπε να οραματιστεί το μέλλον ή να προτρέξει. Γι' αυτό θα ήθελα να τον συγχαρώ για την εξαιρετική αυτή η εργασία, αλλά όπως είπα και άλλοι συνάδελφοι, πολλά λείπουν γιατί τα εγκρίνουμε στο Στρασβούργο μετά την έγκριση, μετά το προσχέδιο. Άρα, μία ερώτηση προς τον Σαλβατόρε. Αυτά που εγκρίναμε στην Ολομέλεια, στην ενδιάμεση έκθεση, προτίθεστε να υποβάλλετε τροπολογίες για να τα επανεισαγάγουμε ή θα το κάνετε εσείς πώς θα συμπεριληφθούν αυτά τα στοιχεία. Ε, εγώ μπορώ να υποβάλω τροπολογίες. Ε, δεν ξέρω αν θα το κάνετε εσείς. Αν το κάνετε, ας μην επικαλύψουμε τη δική σας εργασία. Δύο άλλα σημεία. Συμφωνώ με άλλους προλαλήσαντες. Νομίζω ότι έχουμε αρκετούς μήνες μπροστά μας για να χτενίσουμε ορισμένες συστάσεις. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε και πολλά άλλα. Δεν θα ήθελα να τα δώσω σε λεπτομέρεια, αλλά νομίζω ότι αυτή η έκθεση θα μπορούσε να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες και σε αντίθεση με την ενδιάμεση έκθεση έχουμε καιρό να το κάνουμε αυτό με τροπολογίες και συμβιβασμούς το Σεπτέμβριο. Τέλος, ο Τιμ Κέρκοπ Μίλησε για τους G8 και για τους φόρους και τη φοροδιαφυγή. Θα μπορούσαν να ανακτηθούν πολύ φόροι, το ποσό είναι τεράστιο. Ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας είπε ότι για να λάβουμε πίσω αυτούς τους φόρους θα έπρεπε να συνδέσουμε τις τράπεζες δεδομένων όλων των κρατών μελών. Δηλαδή θα έπρεπε να γίνει αυτός ο κοινός σύνδεσμος. Αυτό τι σημαίνει, ότι λένε οι Βρετανοί ότι θέλουν να συνεργαστούν με τους πάντες και θέλουν συνεργασία και σε διεθνές επίπεδο. Αυτό δεν είχε προϋποθεί. Εάν η Βρετανική κυβέρνηση θέλει να γίνει αυτή η σύνδεση των ε, τραπεζών δεδομένων, τότε θα ισχύσει κάτι τέτοιο και για τα ε, αποτυπώματα DNA, για τα διάφορα μητρώα, αυτοκινητοβιομηχανίας και πολλών άλλων. Αυτό θα πρέπει να το δούμε και σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα, της τράπεζες δεδομένων που υπάρχουν γι' αυτό. Η Επιτροπή μας θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει, ότι ορισμένα κράτη-μέλη αναγνωρίζουν ότι θα πρέπει να μοιραστούν τα στοιχεία που διαθέτουν και όχι να εργαστούν από μόνα τους. Έτσι η έκθεση αυτή ενισχύεται ιδιαίτερα. Η κυρία Μπορσελίνο ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον κύριο Γιακολίνο για την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλε έτσι ώστε να ενσωματώσει σε αυτή την έκθεση τα περισσότερα στοιχεία τα οποία έχουμε προαναφέρει στις διάφορες συζητήσεις, συναντήσεις αλλά και ακροάσεις. Το, ο όγκος είναι εντυπωσιακός. Πολλοί είπαν ότι είναι εκτενής η έκθεση, άλλοι είπαν όμως ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να μιλήσουμε για αυτά τα ε, θέματα, διότι καταβάλαμε κάθε προσπάθεια για να ενσωματώσουμε κάθε δυνατό στοιχείο. Θα ήθελα να υπενθυμίσω κάτι το οποίο θεωρείται δεδομένο. Η έκθεση αυτή δεν είναι μια έκθεση νομοθετικού περιεχομένου. Δηλαδή αυτό που θα ανακύψει είναι συστάσεις και σκέψεις. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι είναι σχηνοτενής αυτή η έκθεση, διότι δεν προτείνουμε, δεν προβάλλουμε μία πρόταση νομοθετικού περιεχομένου. Προτείνουμε τα κράτη-μέλη να ασχοληθούν με θέματα που δεν τα είχαν αποσχολήσει μέχρι τούδε ή τα είχαν απασχολήσει ευκαιριακά και επιφανειακά. Θα πρέπει λοιπόν να ενημερωθούμε για τα τελευταία δεδομένα, ώστε να έχουμε ε, μία βάση εργασίας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιακολίνο για την προσπάθεια που κατέβαλε για να συμπεριλάβει τις προτάσεις όλων. Υπάρχουν ε, θέματα που θα πρέπει να ενισχυθούν, αλλά όλα ενυπάρχουν. Ε, θα ήθελα να πω ότι ως προς τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο ίσως θα ήταν καλύτερα να αφήσουμε αυτή την διευκρίνηση που έχει γίνει στην άκρη. Θα πρέπει να ορίσουμε καλύτερα το πλαίσιο λειτουργίας και όπως είπε η κυρία Φαγιόν, ίσως έχουν εκλείψει ορισμένα στοιχεία. Δηλαδή δεν γίνεται λόγος για οργανωμένο έγκλημα εκτενώς. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ποιος είναι ο μύτος που διέπει το οργανωμένο έγκλημα που ονομάζεται μαφία. Και σήμερα το πρωί είχαμε μία πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση, χωρίς αθρώα προσέλευση, δυστυχώς, όπου τονίσαμε πολλές πτυχές του ζητήματος. Δηλαδή, είπαμε, μιλήσαμε για στοιχεία που πρέπει να αναφερθούν και η επανάληψη δεν είναι κακή στην περίπτωση αυτή. Υπάρχουν και θέματα που έχουν υποτιμηθεί ή αποσιωπηθεί, αλλά εδώ αναφέρονται όλα. Επειδή πρόκειται για τα κατευθυντήριες γραμμές, για όποιον στη συνέχεια θέλει να ασχοληθεί, αυτές υπάρχουν και διαμορφώνονται σαφώς. Δεν ε, υπάρχει πάντα κατακαιρματισμός, δηλαδή έχουμε κάνει έναν απογραφικό κατάλογο των θεμάτων προς διερεύνηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συνεισέφεραν μέσω τροπολογιών και ελπίζω όταν εγκριθεί αυτή η έκθεση να αποτελέσει ορόσημο για μελλοντικές δραστηριότητες. Δηλαδή να πούμε ότι επιτέλους σε αυτή τη θητεία ασχοληθήκαμε με αυτό το ακαθόδε ζήτημα και έτσι αφήνουμε και εμείς το δικό μας ίχνος για τους μεταγενέστερους. Καρόνα. Θα ήθελα ζητήσω συγγνώμη γιατί έφτασα κάπως καθυστερημένα Μπορείτε να, μου πείτε, να μας πείτε στο τέλος ποια είναι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών και ούτω καθεξής δεύτερον. Αφού άκουσα την παρέμβαση της κυρίας Μπορσαλίν, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ. Αλλά θέλω να ξέρω ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτής της έκθεσης και της ενδιάμεσης διότι αν αυτή η έκθεση έχει ως στόχο να ανακεφαλαιώσει μία σημεία, έχει καλός. Εάν έχει στόχο να διευρύνει αυτό το πλαίσιο που μόλις ψηφίσαμε, τότε σημαίνει κάτι το εντελώς διαφορετικό. Τέλος, θα ήθελα να πω τα εξής στον κύριο Γιακολίνο. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ενισχύσουμε το θέμα το οποίο συζητήσαμε και σήμερα το πρωί, επί του οποίου συμφωνούμε όλοι. Δηλαδή το θέμα του οργανωμένου εγκλήματος είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ε, πανάκια όπως το αντιμετωπίζουμε το θέμα της, ε, του οργανωμένου εγκλήματος ως προς τις δραστηριότητες της μαφίας θα πρέπει να μπει ως ξεχωριστό κεφάλαιο. Και ένα τρίτο θέμα είναι ο ρόλος των ε, διαφόρων επιτιδευμάτων δηλαδή δικηγόρων, συμβολεογράφων κλπ. Και συμμετοχή, ενδεχόμενη συμμετοχή συμπεγνία με το οργανωμένο έγκλημα. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν σκόπιμο να υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία και στο τελικό έγγραφο. Ο κύριος Μποργέτσιο. Ευχαριστώ και εγώ δέχομαι τις ε, θετικές παρατηρήσεις και σχόλια που ακούστηκαν και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιακολίνιο για το τιτάνιο έργο, το τιτάνιο έργο του και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να διευρύνω κάπως το πεδίο έτσι ώστε να εμβαθύνουμε κάπως το ζήτημα στο μέτρο του δυνατού. Ελέγχθη ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στη μαφία και το θέμα της χρηματοπιστωτικής, χρηματοοικονομικής μαφίας. Με βάση την πείρα μας, Και επειδή και εγώ είχα συντάξει ένα paper για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, χρειάστηκε να σκεφτώ τα όρια των εργασιών μας. Και γι' αυτό φταίω, φταίμε όλοι ή φταίω και εγώ. Δηλαδή πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το ογκώδες κείμενο του κυρίου Μομπούρ της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης που ασχολήθηκε με τους φορολογικούς παραδείσους. Εμείς μιλάμε για μία επιμέρους εργασία, μιλάμε ε, για την Ιταλική μαφία και δεν ξεκινάμε εκ του μηδενός. Θα πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε ότι τη στιγμή που θα πρέπει να υπάρξει μία ευρωπαϊκή κατεύθυνση για την καταπολέμηση αυτή και τη στιγμή που μιλάμε για μία ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική συντεχνία θα πρέπει να εμβαθύνουμε για να δούμε ποιες είναι οι συναφείς δραστηριότητες και συνεργασία του City του Λονδίνου που είναι κράτος εν κράτη. Και αυτό το λέει η έκθεση αυτή της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε περαιτέρω το όλο ζήτημα. Ο Κάμερον, τον οποίο συμπαθώ και πολιτικά, είπε ότι θα πρέπει να έχουμε επιτάπητος όλα τα στοιχεία. Αν υπάρχει όμως αυτό το νεφέλωμα του ΣΥΤΙ, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι ικανοποιητική η διάθεση αυτών των στοιχείων. Δηλαδή, μας δίνουν τα στοιχεία που επιτρέπει αυτό το νεφέλωμα, δηλαδή σχεδόν τίποτα. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τα παράγωγα που αποτελούν το 70% των παγκοσμίων συναλλαγών του Λονδίνου και για τα παράγωγα δεν μας ε, δίδεται κανένα στοιχείο. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Επιτροπή ΚΡΙΜ και ίσως ε, το ΣΥΤΙ χρηματοδοτεί και ορισμένου πολιτικούς κύκλους προς αυτή την κατεύθυνση. Αν κανείς άλλος δεν θέλει να παρέμβει, πριν δώσω το λόγο στον εισήγητη, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω γιατί ήμουν εισηγήτρια και εγώ μίας έκθεσης που οδήγησε στην δημιουργία αυτής της Επιτροπής με νέα θέματα. Perplessità, e για να μπορέσουν να αρθούν αμφιβολίες, διστάμενες απόψεις και ούτω καθεξής. Ο εισηγητής προσπάθησε να λάβει υπόψη όλες τις θέσεις μέσα στα πλαίσια τη, μιας γενικότερης ε, ε, συμφιλίωσης και λαμβάνοντας υπόψη ότι συμμεριζόμαστε τις απόψεις και των άλλων και εγώ συμφωνώ με αυτά που προείπε η συνάδελφος Μπορσελίνο, ότι δηλαδή πολλές φορές ε, για να μην υπάρχουν αμφιβολίες, για να αρθούν οι αμφιβολίες, ίσως θα, ίσως θα ήταν σκόπιμο να λάβουμε υπόψη και τη λέξη μαφίες, να μην μιλάμε μόνο για οργανωμένο έγκλημα. Ε, η σημερινή ακρόαση ήταν διαφωτιστική και λυπάμαι για τους συναδέλφους που δεν παρευρέθησαν. Ε, δέχομαι αυτό που είπατε εξ αρχής, ότι είχαμε να κάνουμε με 744 τροπολογίες με συντάκτες που πολλές φορές δεν παρευρέθησαν καν στις εργασίες μας. Δηλαδή, εμείς καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να διατρανωθούν συγκεκριμένα μηνύματα και να δώσουμε το στίγμα μας, ενώ δεν υπάρχει αθρώα προσέλευση στις ακροέ, ακροάσεις. Εμείς είχαμε δύο ενότητες, δύο πάνελ δικαστικών και αστυνομικών αρχών που μας είπαν σαφέστατα ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο ανακύπτει από την ανάγκη εναρμόνισης των δικαστικών ε, συστημάτων, αλλά όλα πορεύουν από το γεγονός ότι είτε οι δικαστές ε, είτε οι ανακριτές για να μπορέσουν να διακρίνουν το οργανωμένο έγκλημα χρειάζονται επιπρόσθετα στοιχεία. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κατατρόπωση του οργωμένου εγκλήματος, γιατί χρειάζεται σωρία νομοθετημάτων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εάν θέλουμε να προσπαθήσουμε να κατατροπώσουμε από κοινού το οργανωμένο έγκλημα, μας είπαν σήμερα το πρωί ότι πρέπει να μιλάμε με την ίδια γλώσσα είτε από πλευρά συμμετοχής των ανακριτικών αρχών είτε των δικαστικών να μιλάμε για τα ίδια μέσα. Ε, σήμερα το πρωί μιλήσαμε για γεγονότα και πρακτικές και είδαμε ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνουν μεγάλες κατασχέσεις ε, ναρκωτικών για τη Ιταλία και σε άλλες χώρες υπάρχει η καθυστερημένη σύλληψη, η εκτονιστέρων των σύλληψη, ενώ σε άλλες χώρες όχι. Έτσι, καθυστερούμε και διονγκώνουμε το οργανωμένο έγκλημα, την ουσία του, το περιεχόμενό του. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και αυτήν την ορολογία, γιατί φέτος εργαστήκαμε για να καταστήσουμε σαφές αυτό το μήνυμα. Και για να απαντήσω στον κύριο Καρόνα, η προθεσμία είναι στις 26 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα για την υποβολή τροπολογιών. Αλλά θα το δούμε και στους συντονιστές, διότι οι υπηρεσίες μας είπαν ότι μέχρι τότε δεν θα υπάρχουν, δεν θα έχουμε τις μεταφράσεις, δεν θα έχουμε τη μετάφραση. Θα το δούμε στους συντονιστές αυτό. Αυτή τη στιγμή η προθεσμία είναι 26 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα. Εγώ θα ήθελα πριν δώσω το λόγο στο κύριο Γιακολίνο για να απαντήσει, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και τις ομάδες και θα ήθελα η Επιτροπή να υπερασπίσει με νύχια και με δόντια αυτή την έκθεση έτσι ώστε να βοηθήσουμε τις δικαστικές και ανακριτικές αρχές στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Για την ασφάλεια και τη δημοκρατία, για την ασφάλεια πρωτίστως των πολιτών. Δίνω το λόγο στον κύριο Γιακολίνο για τα τελευταία του σχόλια. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και για την κατανόηση και για την ε, εργασία που ολοκληρώνεται ως προς τις ε, δραστηριότητες αυτές που μας απασχόλησαν εδώ και ένα χρόνο. Ακούσαμε δεκάδες εμπειρογνωμόνων, διαβάσαμε πληθώρα εγγράφων. Πολλοί συνάδελφοι συνέταξαν επιμέρους paper και για την ενδιάμεση έκθεση και για την τελική. Θα ήθελα να εκφράσω ορισμένες σκέψεις ως προς τις παρατηρήσεις που άκουσα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τους φορολογικούς παραδείσους και τουλάχιστον να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα, ε, όπως είπε και ο συνάδελφος Μποργέτζιο. Η Τάνια μας είπε πολύ σωστά ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί εμπιστοσύνη στους, ε, των πολιτών, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλές φορές θα πρέπει να δώσουμε σαφείς κατευθυντήριες γραμμές, δηλαδή σε περίπτωση υποψίας να μην υπάρχει δυνατότητα επανεκλογιμότητας τη στιγμή που έχουν καταδικαστεί ή είναι υπόδικοι. Αναφερθήκατε και στο θέμα της ε, Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι από πλευράς μη Ιταλών συναδέλφων έγινε λόγος για πλήρη αναφορά του οργανωμένου εγκλήματος σαν ξεχωριστή κατηγορία και να μιλάμε και για τη μαφία ξεχωριστά. Εάν θέλουμε όμως να αναφερθούμε και στη μαφία, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ως προς την ε, παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, λάβαμε υπόψη το σημείο 25, τα λάβαμε υπόψη αυτά στο σημείο 25, όπου, όπου γίνεται αναφορά στη... στον ιδιωτικό τομέα και στην παροχή υπηρεσιών ε, μέσω διαδικτύου. Και στο L εννοούμε, επεξηγούμε τι εννοούμε για προμήθειες και παροχή υπηρεσιών. Πρόκειται λοιπόν για τροπολογίες συμβιβασμού που μας απασχόλησαν Λοιπόν, σημείο 25 της ενδιάμεσης έκθεσης και L της τελικής έκθεσης για την ε, τυπολογία αυτών των υπηρεσιών. Εν πάση περιπτώσει είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις και ως προς το θέμα των ε, τυχερών παιχνιδιών. Βεβαίως υπάρχουν υπάρχουν ε, και τα παράνομα παιχνίδια ή τα στημένα παιχνίδια που θα πρέπει να μας απασχολήσουν, απασχολήσουν ξεκινώντας από το ποδόσφαιρο και επεκτηνόμενοι οπουδήποτε. Ο συνάδελφος Σοντεγκάρντα αναφέρθηκε σε ορισμένες ε, τροπολογίες που σχετίζονται με το, τη συμπλήρωση αυτής της εργασίας. Θα ήθελα να πω ότι και για μένα το έργο αυτό είναι τιτάνιο. Ο κύριος Αλμπρέχτ μίλησε για τις πολιτικές προτεραιότητες αυτής της έκθεσης Συμβαδίζω με την κυρία Μπορσελίνο, η οποία είπε ότι άλλοι θεωρούν ότι η έκθεση αυτή είναι πλημμυρίδα και άλλοι τη θεωρούν μία σταγόνα και μόνο στον ωκεανό. Ε, όμως, θα έχουμε 27 σελίδες, ενώ η ενδιάμεση έκθεση ε, είχε 38. Προσπαθώ λοιπόν να δώσω τις βασικές κατευθυντηρίες γραμμές. Και στο σημείο 1 της τελικής έκθεσης όταν αναφέρεται ότι επαναλαμβάνονται τα δεδομένα της ενδιάμεσης έκθεσης με ψήφισμα της 11ης 13. Το παρόν ψήφισμα προτίθεται να τις επιβεβαιώσει, τις διαπιστώσεις αυτές δηλαδή, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητός. Όλα αυτά τα οποία εγκρίθηκαν από την ενδιάμεση, στην ενδιάμεση έκθεση ισχύουν. Αυτό το λέω και για τον Μπιλ. Ό,τι έχει εγκριθεί από την ενδιάμεση έκθεση βεβαίως ε, ενυπάρχει. Αν και δεν αναφέρεται ρητός. Ο συνάδελφος Άλμπρεχτ μιλά για εναρμόνιση των ε, διατάξεων νομοθετικού περιεχομένου ε, σας προτείνω να διαβάσετε το, την έκθεση γιατί υπάρχουν πολλά από αυτά τα στοιχεία τα οποία εσείς θεωρείτε απόντα μιλώντας και για την συνεργασία δικαστικών και αστυνομικών αρχών και την ανάγκη συμφωνιών συνεργασίας με τρίτες χώρες μέσα στα πλαίσια πληροφοριών που χρειάζονται οι ανακριτικές αρχές για να μπορέσουν να στεφτούν από επιτυχία το εγχείρημά τους. Ο Μπιλ αναφέρθηκε στην απέτηση αυτής της διάθεσης πληροφοριών. και στην Ολομέλεια υπήρξαν τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση που εγκρίθηκαν. Είμαι στη διάθεσή σας και θα είμαι και στους συντονιστές για να σας δώσω άλλες πληροφορίες αν τις θέλετε. Κυρία Μπορσελίνο, αναφερθήκατε για το ότι δεν είναι μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου, πρόκειται για ένα πολιτικό στίγμα από τη δική μας πλευρά. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ολοκληρωμένα και το τελικό και το ενδιάμεσο κείμενο. Υπάρχει ένα σαφές περιεχόμενο και όλα τα επιμέρους στοιχεία που επιβάλλονται. Εάν κρίνετε ότι κάτι λείπει, να το υποβάλλετε σας παρακαλώ υπομορφή τροπολογίες ως προς τη μαφία. Είπε πολύ σωστά και η κυρία Μπορσελίνο ότι θα πρέπει να αναφέρεται ρητά κάτι το οποίο θα λάβουμε υπόψη και στις τροπολογίες. Βεβαίως εδώ μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα τα οποία τροφοδοτείται από άλλα εγκληματικά συστήματα και υποβοηθάται από την υπέρογγη γραφειοκρατία. Γι' αυτό χρειάζονται μεταρρυθμίσεις ιδιαίτερα σε ορισμένε χώρες. Το θέμα της μαφίας, της διαφθοράς και της ανακύκλωσης είναι ένα θέμα που αφορά όλα τα κράτη-μέλη. Πρόκειται για διεθνικά εγκλήματα και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε και το σύστημα της ΕΚΟ-ΜΑΦΙΑ. Το είδαμε κύριε Καρόνα αυτό όταν αναφερθήκαμε και στα επιτιδεύματα, ε, δηλαδή λογιστές, ε, εμπορικά επιμελητήρια, συμβολεογράφοι, δικηγόροι. Μιλάμε για τις συστάσεις που επιβάλλονται στο σημείο 52. Στο σημείο 52 υπάρχει η αναφορά των επιτιδευμάτων όπου μιλάμε για παράνομες δραστηριότητες και συναλλαγές καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο συνάδελφος Καρών Αναφέρθηκε και στα αδικήματα κατά του περιβάλλοντος, ενώ ο συνάδελφος Βοργέσιο αναφέρθηκε ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η μαφία τροφοδοτείται και από το οικονομικό έγκλημα και από την αγορά των παραγόγων Μιλήσαμε για ένα 70% των δραστηριοτήτων του City. Θα λάβουμε υπόψη λοιπόν τις παρατηρήσεις και τη συνεισφορά της Πρόεδρου Αλφάνου, την οποία ευχαριστώ, καθώς και όλους εσάς για να δούμε αυτή την κρίσιμη φάση διασύνδεσης της ε, ενδιάμεσης έκθεσης με αυτήν. Δηλαδή μετά από την βροχή των 744 τροπολογιών έχουμε φτάσει σε μία ανασυγκρότηση της σκέψης μας με 77 τροπολογίες συμβιβασμού. Άρα, μιλήσαμε και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για τους μάρτυρες, για την αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού εγκλήματος, για το διεθνικό χαρακτήρα αυτών των εγκλημάτων, όπου χρειάζεται ευρεία συμμετοχή όλων των κρατών μελών και των τρίτων χωρών. Πιστεύω ότι αυτή η εργασία μπορεί να βελτιωθεί, αλλά τα ουσιώδη στοιχεία έχουν αναφερθεί και στις δύο εκθέσεις. Θα δούμε μέχρι τις 26 Ιουνίου πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε όλα αυτά τα επιμέρους στοιχεία στις 26 της 5 το απόγευμα πρέπει να υποβληθούν τυχόν τροπολογίες. Και στη συνέχεια θα προβούμε σε μία συγκεφαλαίωση έτσι ώστε οι τελικοί αποδέκτες αυτού του εγγράφου να γνωρίσουν τις πολιτικές προτεραιότητες που έχουμε εμείς θέσει. πιστεύοντας ότι στο εγγύς μέλλον θα φτάσουμε και στην Τραπεζική Ένωση, η οποία θα είναι χρήσιμη και για τις δικές μας υποθέσεις. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστούμε κύριε Γιακολίνο. Εάν δεν υπάρχουν άλλες ε, παρατηρήσεις από τους συναδέλφους, φαίνεται πως όχι. Ο Μπίλ. Μια στιγμή, να διευκρινίσουμε κάτι. Μπορούμε εμεί να κάνουμε διάμεση έκθεση και τελική έκθεση, άρα είμαστε και ένα μοναδικό φαινόμενο. Οι άλλε επιτροπέ δεν το κάνουν αυτό. Τι λένε λοιπόν τα άρθρα του καταστατικού. Πράγματα τα οποία ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην ενδιάμεση έκθεση, αλλά δεν περιλαμβάνονται στην τελική. Πρέπει να τα επαναλάβουμε ή θα διανεμηθεί η ενδιάμεση έκθεση μαζί με τα τελικά μας συμπεράσματα. Για μένα αυτό είναι ένα κενό που αφήνει ο κανονισμός. Τι, μπορεί, τι θα συμβεί εδώ. Ήδη το είπε, πρόκειται για το άρθρο υπαριθμών 1. Πιλ στο άρθρο υπαριθμών 1 της τελικής έκθεσης υπάρχει μια πρόβλεψη η οποία ενσωματώνει ό,τι εν υπάρχει στην ενδιάμεση έκθεση. Το περισσώζει, αν θέλετε. Δηλαδή εγκρίναμε την ενδιάμεση, αλλά δεν θέλουμε να επαναλάβουμε τα ίδια. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μία άσκηση ορθολογισμού και περιλαμβάνουμε όλα τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται, χωρίς να προδικάζουμε το μέλλον. Για λόγους οικονομίας χώρου, δηλαδή, θεωρήσαμε ότι ότι θα πρέπει με αυτή τη ρήτρα διασφάλισης ε, να θεωρήσουμε ότι περιλαμβάνουμε όλα τα προγενέστερα. Θα το δούμε στους συντονιστές βεβαίως, αν υπάρχουν ε, κενά. Για να ορίσουμε και τον ε, τρόπο προώθησης της όλης διαδικασίας. Νιούτον Ευχαριστώ Σαλβατόρε. Διάβασα την έκθεση, βεβαίως και την, παράγραφο, την πρώτη παράγραφο του άρθρου πρώτο. Ευχαριστώ για την εξήγησή σου. Τώρα, σε ό,τι προβλέπει ο κανονισμός του Κοινοβουλίου, δεν υπάρχει προηγούμενο, αναφερόμαστε, δηλαδή παραπέμπουμε σε προηγούμενο έγγραφο και λέμε ότι αυτό είναι απόφαση που έχει λάβει το Κοινοβούλιο. Ίσως κανείς από εμά που είμαστε παρόντες τώρα να μην μπορεί να απαντήσει. Είναι όμως επαρκής η διαβεβαίωση που δίνει ο Σαλβατόρε ή απαιτείται να επαναλάβουμε τα συμπεράσματά μας στην τελική έκθεση. Δεν θέλω δηλαδή να παραλυφθούν κάποια πράγματα που είναι πολύ σημαντικά. Πρόεδρος, όσον αφορά τις ανησυχίες σου, δεν υπάρχει κανένας τέτοιος κανονισμός. Τη στιγμή που η πρώτη έκθεση, η διάμεση έκθεση ενεκρίθη την τρίτη, τη στιγμή λοιπόν που εγκρίνεται από την Ολομέλη, αποτελεί μια εγκεκριμένη πράξη. Όταν εγκριθεί και η τελική έκθεση, εάν εγκριθεί με, την πλειοψηφία, εάν ε, ε αν υπάρξει έγκριση με πλειοψηφία, τότε θεωρείται κάτι το ευρέως αποδεκτό αλλά μέσα στα πλαίσια της σύνταξης ε, μπορείτε, αν θέλετε, με τροπολογίες ε, να ενισχύσετε το κείμενο. Θα ήθελα να πω στο Bill ότι στο τελικό κείμενο θα αναφερθούμε σαφώς στην ε, ενδιάμεση έκθεση που εγκρίναμε. Δηλαδή, θα πούμε λαμβάνοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση υπαριθμών τάδε κλπ. κλπ. Θα αναφερθούμε δηλαδή στην ε, τελική έκθεση ε, για να ενισχύσουμε αυτό ακριβώς που προανέφερε η Πρόεδρος. Ωραία, νομίζω ότι το θέμα αυτό ε, το είδαμε επαρκώς. Λοιπόν, στις 26 Ιουνίου μέχρι τις 5 το απόγευμα πρέπει να έχετε υποβάλει τροπολογίες και σε λίγα λεπτά αρχίζει η συνάντηση των συντονιστών, δηλαδή στις 4.30 ακριβώς. Σας ευχαριστώ και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.